przewodniczący! Καλημέρα σας κυρίε και κύριοι, παρακαλώ λάβετε θέσεις. Θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω στην ε, Σύνοδο της Ολομέλειας. Θα ήθελα καταρχήν να σας ε, κοινοποιήσω δύο λυπηρές πληροφορίες. Χθες στη, Φλωρέδη, ε, στη κάποιος ε, πυροβόλησε δύο ανθρώπους για ρατσιστικούς λόγους και για μια ακόμη φορά έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι που ήθελαν να ζήσουν και να εργαστούν στην Ευρώπη. Αυτό είναι εξαιρετικά λυπηρό και σίγουρα θα πρέπει αποφασιστικά να μην φυστούμε προσπαθειών για να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε ε, δραστηριότητα